της Επιτροπής όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη συντάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και δίνω το λόγο στην κυρία Τάισεν. Ευχαριστώ ξανά κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας πριν από ένα χρόνο, θέσαμε την κοινωνική δικαιοσύνη στο επίκεντρο της δουλειάς μας. Και σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Ο, τη διαφορά 40% όσον αφορά τη συντάξη με βάση το φύλλο, η έμφυλη αυτή διαφορά είναι απαράδεκτη. Από 4 μέχρι 46% ποικίλει διαφορά σε διάφορες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι σαφές ότι οι πολιτικές κάνουν τη διαφορά. Θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε και να επιδιώξουμε ίσες ευκαιρίες και σχετικές πολιτικές να εφαρμόσουμε σε διάφορους τομείς. Πολύ πριν φτάσουν οι άνθρωποι στην ηλικία συνταξιοδότησης, ήδη το κάνουμε αυτό και θα αναλάβω περαιτέρω σχετικές δράσεις. Πριν το τέλος ενεστώτος έτους θα παρουσιάσουμε στατηγικές υποχρεώσεις για την ισότητα των φύλων. Θέλουμε να καθορίσουμε τη γενική βάση για ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Στόχος τους η βελτίωση ισότητας των φύλων. Θα αντιμετωπίσουμε και τα αίτια της διαφοράς όσον αφορά τις συντάξεις. Όπως ξέρετε, το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μία νέα αρχή για τους εργαζομένους ε, ε, γονείς και τους διάφορους περιθάλποντες ε, και θέλουμε να εξισορροπήσουμε τα δύο φύλλα και θέλουμε καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Μια νέα προσέγγιση θα είναι επωφελής και για τους εργαζόμενους γονείς και τους άλλους που περιθάλπουν άτομα στο σπίτι τους ε, για να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις τους και θα μπορούν και οι γυναίκες να ε, μπορούν να συμμετέχουν καλύτερα στην αγορά εργασίας. Θα γίνεται καλύτερος επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών και θα ε, τονώσουμε την ισότητα των φύλων. Η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και η ανοιχτή δημόσια διαβούλευση από αυτών ήδη δρομολογήθηκαν και ξεκίνησαν. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις διευθετήσεις για άδειες Θέλουμε να προωθήσουμε ευέλικτες διευθετήσεις για την εργασία και υπηρεσίες ε, φροντίδας ποιοτικέ. και να μην ε, θα πρέπει να υπάρχουν και κίνητρα στα διάφορα ε, συστήματα, στα ευεργετήματα που δίνονται στις γυναίκες. Θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στην αγορά εργασίας οι γυναίκες και να μην επιβαρύνονται λόγω των καθηκόντων τους ως μητέρες. Θα πρέπει λοιπόν να καλύψουμε τα προβλήματα όσον αφορά τα δικαιώματα συνταξιοδοσία, ε, που υπάρχουν οι διαφορέ που τάξουν μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα αναλάβουμε δράσεις για διαμόρφωση πολιτική και για ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη διαφορά αμοιβών, την έμφυλη διαφορά. Το 2016 θα διαθέσουμε 4 εκατομμύρια ευρώ, θα τα δώσουμε στα κράτη-μέλη για ευαισθητοποίηση όσον αφορά την έμφυλη διαφορά στον αφορά τη συντάξει και τους λόγους που ε, οδηγούν σε αυτή την ε, διαφορά. Πώς προσμετράμε, προσμετράτε η διαφορά. Παρακολουθούμε το θέμα όσον αφορά τις συντάξεις και κατά πόσο είναι επαρκείς οι συντάξεις και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των συντάξεων. Η Eurostat τακτικά θα επικαιροποιεί τα στοιχεία όσον αφορά το θέμα αυτό. Θα συνεχίσουμε το έργο μας. Θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη στις Επιτροπές Απασχόλησης Προστασίας των Εργαζομένων να δούμε ποια μεθοδολογία εφαρμόζεται και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Θα χρησιμοποιήσουμε βεβαίως διάφορες εκτιμήσεις και δείκτες διαφορών, εμφύλων διαφορών στο έργο που θα κάνουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα εξετάσουμε άλλους βασικούς δείκτες όπως και τι γίνεται με τους φτωχούς ηλικιωμένους, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των φύλων στοιχεία για τη διαφορά των συντάξεων προέρχονται από δίκτυ που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξέτασαν οι εμπειρογνώμονε για την ισότητα των φύλων το δίκτυ και θέλουν να αναπτύξουν το δίκτυ. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία εδράζονται επί βελτιωμένη μεθοδολογία. Εισήχθησαν στην έκθεση του 2015 για την επάρκεια των συντάξεων. Η αρμόδια επιτροπή για τι συντάξει ανέπτυξε το δίκτυ. Προσμετρούμε πώς οι πρώτερες διαφορές, οι έμφυλες, στην απασχόληση, ώρες εργασίας κλπ. και διάρκεια καριέρας, πώς αυτά επηρέασαν τις διαφορές στις συντάξεις και στα δικαιώματα τα συνταξιωτικά. Σε κάποιο βαθμό τα συνταξιωτικά συστήματα μπορούν να μειώσουν το πλήρη αντίκτυπο των διαφορών των παλαιών, των προηγουμένων όσον αφορά την απασχόληση ελάχιστη σύνταξη και λοιπά, ε, δικαιώματα συνταξιωτικά και να δώσουμε περισσότερη προστασία στις γυναίκες όσον αφορά της συντάξεις. Και χωρίς αυτά τα συστήματα περαιτέρω προστασίας, τα κενά και έκθεση στους κινδύνους για να γίνουν φτωχές οι γυναίκες θα ήταν μεγαλύτερη η κίνδυνη. Πέρα από τη βελτίωση των φύλων και την απασχόληση των γυναικών, θέλουμε να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε και τα μέτρα διαφύλαξης και προστασία των γυναικών. κλείνοντα θετικά, να τονίσω ότι λόγω της συνεχούς αύξησης τη απασχόληση των γυναικών στα περισσότερα κράτη-μέλη τις τελευταίες τρει δεκαετίε, οι μεγαλύτερε έμφυλες διαφορές μειώνονται και καμιά φορά κατά... σε πολύ σημαντικό βαθμό. Όμω, αν δεν εκριζώσουμε τις έμφυλες διαφορές στην απασχόληση θα συνεχίσουν να εμφανίζονται οι διαφορές και στις συντάξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να καλύπτει τις διαφορές στις συντάξεις, αλλά θα εντατικοποιήσει και περαιτέρω τις προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε τώρα στους αγορητές εκ μέρους των ομάδων για το ΕΛΚ για 1,5 λεπτό. Ανιέσκα Κοζιώσκα Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η κατάσταση οι γυναίκες ε, να μην έχουν αξιοπρεπή σύνταξη είναι άδικη. Έτσι λοιπόν ε, σας ευχαριστώ για όλα όσα είπατε. Εντάξει, μεταξύ των δύο φίλων και σας ευχαριστώ και για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε και που θα αναλάβετε και στο μέλλον γιατί το χάσμα στις συντάξεις ε, μεταξύ των δύο φίλων είναι πολύ μεγάλη αδικία, ιδίως ε, για τις γυναίκες. Και βλέπουμε ότι έχουμε κάποιους συσσωρευμένους δείκτες. Φυσικά θα είναι χρήσιμο για μας να κάνουμε κάτι για να πετύχουμε μεγαλύτερη ισότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να δούμε τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτό το χάσμα στις συντάξεις και όχι μόνο τα συμπτώματα. Φυσικά αυτό έχει να κάνει και με τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, σε πόσο καιρό έχουν δουλέψει και τις εισφορές τους. Όπως είπα, θα πρέπει να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασία και αν θέλουμε να έχουμε υψηλέ συντάξει για τι γυναίκε, θα πρέπει να καταστήσουμε δυνατό να μπορούν να αποκτήσουν οι γυναίκε τέτοια σύνταξη δεν είναι μόνο θέμα ισορροπίας ε, στην εργασιακή ζωή, αλλά θα πρέπει να δούμε και το θέμα της εκπαίδευσης και άλλες πτυχές, έτσι ώστε να μην ε, αποκόβονται οι γυναίκες, να μην διαχωρίζονται από την αγορά εργασίας. Επομένως, οποιαδήποτε στρατηγική αναπτυχθεί, θα είναι κάτι καλό. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί όλα τα κράτη-μέλη και φυσικά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκ μέρου των Σοσιαλιστών, η συνάδελφο Γιούτα Στάινρουκ για 1,5 λεπτό. Ναι. ναι, το γεγονό ότι το φύλλο καθορίζει την ε, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις συνθήκες εργασία και κυρίω την αμοιβή και οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κερδίζουν 16% ε, λιγότερο από τους άντρες και αυτό βεβαίως αντανακλάται στις ε, συντάξεις αργότερα. Και η Επιτροπή, είπατε κυρία Τάισεν, προτίθεται να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Η φροντίδα των παιδιών, λέτε, θα βελτιωθεί και οι άντρες θα έχουν περισσότερα κίνητρα να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο. Όλα αυτά είναι ωραία, αλλά δεν επιλύουν το βασικό πρόβλημα που είναι οι μισθολογικές διαφορές, τις οποίες θα πρέπει να εξαλείψουμε και να επιφέρουμε αλλαγές. Χρειαζόμαστε δεσμευτικά προγράμματα για ίση αντιμετώπιση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στον χώρο εργασίας ε, που θα πρέπει να είναι απολύτως υποχρεωτικά και δεσμευτικά. Ε, λέτε ότι θέλετε να συλλέξετε δεδομένα για το χάσμα μεταξύ των ε, φύλων γιατί και μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούν να αμβλυνθούν οι διαφορές της αποδοχές. Διακόπτεται. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα για τους φιλελεύθερους, η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Η, τα δεδομένα για το χάσμα πραγματικά είναι ε, σημαντικά. Ε, στη χώρα μου είναι 40% και το χάσμα για τις συντάξεις είναι και πάλι 40%. Ε, αυτές είναι οι σοκαριστικές ε, στατιστικές και τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσουμε εδώ είναι τα εξή. Πώς μπορούμε να μικρύνουμε αυτό το χάσμα και δεύτερον τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να εξασφαλίσουμε συντάξει των ε, ανέργων να γίνουν βιώσιμες. Χαίρομαι που αναφέρατε ορισμένες πιθανές λύσεις για παράδειγμα την, τη συντάξη για τους επιζώντες. Επίσης αναφέρατε ελάχιστε συντάξεις ή ελάχιστε αποδοχές. Και υποστηρίζω απολύτως αυτές τις προτάσεις. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Προηγουμένως συζητήσαμε για τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Βεβαίως θα πρέπει να τηρηθούν αυτές οι συνθήκες και να υπάρχουν ευέλικτες διαθετήσεις όσον αφορά το ωράριο, ώστε οι άνθρωποι που επιθυμούν να εργαστούν να μπορούν να το κάνουν όσον αφορά την ε, αποχή από την εργασία λόγω νόσου. Ε, θα πρέπει να απαντηθεί ένα θεμελιώδες ερώτημα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποδεκτό αυτοί οι οποίοι απέχουν από την εργασία για να φροντίζουν αυτούς που χρήζουν ε, φροντίδας να απειλούνται από ενεργεία και φτώχεια. Κατά την άποψή μου αυτό είναι απαράδεκτο γιατί τα συστήματα υγείας θα καταρρεύσουν χωρίς την ε, βοήθεια αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό ε, θα πρέπει να εντάξουμε τη φροντίδα και την ανάληψη ευθύνης ήδη εντός των ασφαλιστικών ε, συστημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Μπόιλαν. Ευχαριστώ. Η διαφορά συνταξιοδοτική αυξήθηκε στην Ιρλανδία μετά την οικονομική κρίση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πολλέ γυναίκε δεν μπορούν να έχουν οικονομική ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια που φέρνει αυτή όταν συνταξιοδοτούνται. Ξέρουμε ότι η έμφυλη διαφορά είναι σωρευτική σημαντικό αποτέλεσμα παραγόντων συμπεριλαμβανομένης και της διαφοράς στις αμοιβέ. Πρέπει να αναγνωρίσουμε όταν μιλάμε για προληπτικά μέτρα και αντιμετώπιση των εμφύλων διαφορών όσον αφορά συντάξει, ότι και οι πολιτικέ λιτότητα επιδεινώνουν το πρόβλημα και δεν το μειώνουν. Ε, η εφαρμογή, η πολιτικών που εφάρμοσαν οι κυβερνήσει τη Ιρλανδία από το 2008 και μετά επιδίνωσαν την κατάσταση τη γυναίκα στην Ιρλανδία. Η κυβέρνηση μείωσε τις, τα συντεξιωτικά δικαιώματα για του εργαζόμενου στο δημόσιο τομέα και σε συγκεκριμένου τομεί που ε, είναι οι γυναίκε περισσότερε, όπω είναι οι νοσοκόμε και ε, τομέα διδασκαλία. Μειώσανε του μισθού και τι συντάξει του. Είμαστε, έχουμε, τα, έχουμε τα ψηλότερα επίπεδα χαμηλά αμοιβωμένων εργασι, θέσεων εργασία ε, μετά τη ΣΥΠΑ. Και πάνω από 60% από αυτέ τι ε, θέσει είναι στα χέρια γυναικών. Και βλέπουμε παρόμοιε τάσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω και το κόστο για την φροντίδα των παιδιών είναι υψηλό στον κόσμο. Πάνω από 40% του μέση της μέσης αμοιβή στην Ιρλανδία. Και έτσι εξαιρούνται οι γυναίκε. Δεν μπορούν να, να συμμετάσχουν στην παραγωγική οικονομία ή πρέπει να βρουν θέσει εργασία επισφαλή. Και δεν μπορούν να συμβάλλουν στα συνταξιωτικά συστήματα. Πολλά βήματα μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετώπισουμε την έμφυλη διαφορά συντάξει, αλλά θα πρέπει να παραδεχτούμε πρώτα απ' όλα ότι έχει καταστροφικό αντίκτυπο η πολιτική τη λιτότητα η οποία εφαρμόζεται. Είναι καταστροφική για τι γυναίκε, πρέπει να αντιστραφούν τα μέτρα λιτότητα. Ευχαριστώ για μισή λεπτό, Μαρία Ρένα. Ah, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για όσα μας είπατε. Είναι αλήθεια ότι το χάσμα στις ε, συντάξεις δεν είναι κάτι που συμβαίνει στα 65 έτη, είναι κάτι που οικοδομείται καθ' όλη τη σταδιοδρομία, ίσως και πριν τη σταδιοδρομία, γιατί στις γυναίκες ε, μας ε, έχουν αποδώσει κάποιους ρόλους, ήδη τη στιγμή που διαλέγουμε τις σπουδέ μας, γιατί βλέπουμε όσο λιγότερα προσόντα έχει κάποιος, τόσο μεγαλύτερο είναι το χάσμα στις συντάξεις. Επίσης, αναφερθήκατε και Τη διακρίσεις στην αγορά εργασία υπάρχει και το θέμα τη ημερική απασχόληση που δεν αντισταθμίζεται όταν υπολογίζεται η σύνταξη. Υπάρχει στο διοδρομέα, υπάρχει το θέμα τη μητρότητα με ε, τι γονικέ άδειε και την άδεια μητρότητα. Υπάρχει και η ανισότητα ε, γιατί δεν έχουν πρόσβαση, την ίδια προσβασία οι άντρε. Επίση, υπάρχει το θέμα τη μη συμφιλίωση ιδιωτική, ε, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Επίση, ε, υπάρχει και το θέμα ε, των χαμηλόμιστων επαγγελμάτων, αλλά και στο, στον κλάδο των γυναικών δεν υπάρχουν συντάξει δεύτερου και τρίτου πυλώνα. Έτσι, λοιπόν, όλα αυτά μα οδηγούν στην φτωχοποίηση των γυναικών. Αναφέρατε διάφορα στοιχεία. Εγώ αναφέρω και άλλα που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο στα πλαίσια του σχεδίου δύο ισότητα των δύο φύλων. Θα επανέλθω με το θέμα της γονικής άδεια, την άδεια που θα πρέπει να πληρώνονται, τις υπηρεσίε της οικογένειας που θα πρέπει να είναι προσωπισμένες και ένα πρώτο πυλώνα συντάξει που θα πρέπει να τροφοδοτείται σωστά. Ε, σήμερα βλέπουμε στην Ευρώπη ότι υπάρχει συρρήκνωση του πρώτου πυλώνα της σύνταξης. Εδώ ολοκληρώνουμε τον κατάλογο των μενητών. Ερχόμαστε στο Catch the Eye. Κυρία Ροντρίγκε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι αγρότησες ε, που εργάζονται στις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη είχαν και συνεχίζουν να έχουν πολλές δυσκολίες για να ε, πάρουν ε, σύνταξη και να δώσουν εισφορά στην κοινωνική ασφάλιση. Αυτό για νομικούς λόγους, για οικονομικούς αλλά και πολιτιστικούς λόγους. Αλλά όλα αυτά έχουν βάση ε, στο ότι οι γυναίκες υφιστάμεθα διακρίσεις. Στα τέλη του 20ου αιώνα υπήρχαν σημαντικοί αγώνες από τις αγρότησες στην Αυστρία για να πετύχουν το δικαίωμα στη συνταξιοδότηση και επίσης και από τις αγρότες στη Γαλλικία που ήταν παντρεμένες με άνδρες που είχαν άλλα επαγγελματία και καθώς κέρδιζαν περισσότερο από αυτές τους ε, αρνούνταν το δικαίωμα να πληρώνουν την κοινωνική ασφάλιση. Έτσι λοιπόν αυτό σημαίνει στο να έχουν μικρότερε συντάξει σήμερα οι αγρότες από του αγρότε. Σα ζητώ κύριε Επίτροπε όταν αναλύσετε αυτέ τι προτεραιότητε για τη μείωση του χάσματος στι συντάξει, να λάβετε υπόψη και τι αγρότησε. και παρακαλώ αφήστε με να ολοκληρώσω. Αυτό περνά από την πλήρη αναγνώριση των δικαιωμάτων των αγροτησών. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό. Δεν το για Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε να καταπολεμήσουμε τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών επί έτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα όμως υπάρχει δραματικό ε, πρόβλημα με τη διαφορά στις συντάξεις. Αν δείτε τις διαφορές που υπάρχουν στους μισθούς, περίπου 13% στη συντάξη διαφορά είναι μεγαλύτερη. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε κρίση. Και για πολλά χρόνια κατανοήσαμε ότι η πηγή της διαφοράς των συντάξεων είναι η μη ισότιμη αντιμετώπιση στην αγορά εργασίας. Γνωρίζουμε ότι έχουμε στατηγική την Ευρώπη για το 2020 και ότι πρέπει να προοδεύσουμε στον τομέα της διάκρισης κατά των γυναικών. Πολύ συχνά οι γυναίκες εργάζονται σε χειρότερες συνθήκες και αν δείτε τι γίνεται με τι γυναίκε, μία στι τέσσερι ποτέ δεν είχε μία επίσημη θέση εργασία. Και έχουν πρόβλημα αυτέ οι γυναίκε όσον αφορά τα συνταξιδωτικά του δικαιώματα. Προφανώ αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε μία κρίση που επιδεινώνεται στην περίπτωση των διαζευμένων γυναικών. Ευχαριστώ. Τελευταία ομιλήτρια για, για ένα λεπτό. Κυρία Ζούμπερ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν καλύτερα προληπτικά μέτρα για να απεθύγουμε τη διάκριση μεταξύ των δύο φύλων με το να ε, δώσουμε τέλος ε, στο χάσμα αυτό και γι' αυτό πρέπει να σεβαστούμε τις συλλογικέ συμβάσεις, να αποφύγουμε να έχουμε ατομική διαπραγμάτευση. Ε, οι εργαζόμενες δεν έχουν τρόπο να καταγγείλουν ε, αυτές τις διακρίσεις. Ε, θα πρέπει να έχουμε πιο κατάλληλα μέσα και θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στις επιχειρήσεις που δεν σέβονται την νομοθεσία, να πρέπει να περασπίσουμε τα δικαιώματα της μητρότητας έτσι ώστε να μην ζημιώνονται οι γυναίκες ε, στις συντάξεις επειδή κατά την εργασική του ζωή ήταν και μητέρες. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα αλλά και οι εφαρμογή τους ε, μαζί με το να έχουμε δημόσια καθολικά και αλληλέγγυα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης θα ε, εγγυηθούν ε, μια αξιοπρεπή σύνταξη για τις γυναίκες. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνοντας θα πάρει πάλι η Επίτροπος κυρία Τάισεν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την υποστήριξη που μου δώσατε εδώ, γιατί πραγματικά είναι αδιανόητο να υπάρχει τέτοιου είδου ε, χάσμα της τάξης του 40%. Και ε, νομίζω ότι θα πρέπει από κοινού να επικεντρωθούμε σε αυτό το έργο. Πώς διαμορφώνει τι αδυναμίες των γυναικών, κάτω από ποιες συνθήκες εργάζονται οι γυναίκες. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις προϋποθέσεις και το βασικό κανόνα ότι θα πρέπει η ίδια εργασία να μείβεται με ίσες αποδοχές. Δεύτερο σημείο, οι ρυθμίσεις για τις συντάξεις και τα ίδια τα συνταξιοδοτικά συστήματα οι ειδικέ προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν εδώ ε, ε, πώς, τι είδου διορθώσεις θα μπορούσαμε να επιφέρουμε στα συστήματα των συντάξεων. Όπως είναι σωστό ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το δεύτερο πυλώνα και είναι ξεκάθαρα νομίζω στη δική μας προσέγγιση ότι δεν θέλουμε μόνο εφικτές ε, ε, συντάξεις αλλά και επαρκείς ε, συντάξεις, δηλαδή συντάξεις που να επιτρέπουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Γι' αυτό θα πρέπει να διευρυνθεί αυτός ο δεύτερος ο πυλώνας και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την διάσταση του φίλου και εκείνους τους τομείς που πρωτίστως απασχολούνται γυναίκες. Μιλήσ... Ακούσαμε για μία πρόταση σε σχέση με την άδεια μητρότητας ε, η οποία ε, επί του παρόντος έχει αποσυρθεί αλλά νομίζω ότι και εδώ θα μπορούσαμε να επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Τάισεν.